Αναλαμβάνουμε, συνάδελφοι, ότι υπάρχουν ψηφοφορίες και σε άλλη επιτροπή. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Okay, colleagues, take... Καθίστε παρακαλώ. Ξεκινάμε με την ψηφοφορία. Καθίστε. Υπάρχουν και άλλες ψηφοφορίες σε άλλες επιτροπές. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε τις άλλες ψηφοφορίες. Ε, θα είναι για την προσ για την πρόταση για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Η Τάνια Φαγιών είναι η συγγήτρια. Θέλει να πάρει το λόγο η συγγήτρια, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα απλά να πω μερικά λόγια για τις συμβιβαστικέ ε, στην έκθεση που θα ψηφίσουμε απόψε. Γνωρίζετε πόσο σημαντική ήταν η, η, η, και πόσο αυτοί οι ελάχιστα ιστορικά σύνορα έχουν ε, αλλάξει τα πράγματα. Με τις συμβιβαστικέ ζητάμε ε, μέγιστο, ε, μέγιστη προθεσμία ενός έτου. Αυτό συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο στο θέμα αυτό και προτείνω ε, επιπρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες για το πώς και πότε αυτοί οι έλεγχοι εσωτερικών συνόρων μπορούν να εισαχθούν και να διατηρηθούν. Αυτές οι δικλείδες είναι για να ε, ενισχύσουν τις δικλείδες που έχει προτείνει η Κομισιόν και οι συμβαστικές ε, ανακλούν μια ισορροπημένη άποψη και αποτελούν βάση για ε, διαπραγματεύσεις σε τριμερή διάλογο, έτσι ώστε να μην παρατείνουμε τους εσωτερικού ε, ελέγχους στα σύνορα και να δούμε για πόσο καιρό μπορούν να εισαχθούν αυτοί οι εσωτερικοί ε, έλεγχοι. Θέλω να στηρίξετε όλες τις συμβιβαστικέ και την έκθεση, συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ σαφή η συγγήτρια σε σχέση με τις συμβιβαστικέ τροπολογίες. Ξεκινάμε λοιπόν για, με τη συμβιβαστική 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι διαδικαστικό, κύριε Αλμάρη. Ναι. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία και μετά θα πάρουμε το διαδικαστικό. Θα ολοκληρωθεί πρώτα η ψηφοφορία, παρακαλώ. Να ολοκληρωθεί πρώτα. Έχουμε την συμβιβαστική τροπολογία 14. Ήμασταν στη μέση της ψηφοφορίας, πέρα της ψηφοφορίας. Δεν λειτουργεί η κάρτα μου. Ήταν για αυτό που είχατε ζητήσει το λόγο. Όχι, δεν ήταν για αυτό. <laughs> Sorry, it doesn't work. Monica. Okay, Monica, do you have a point of order just before I, I get? I try it again. No, it's okay. It's okay. No, it's okay. Τώρα λειτουργεί η κάρτα. Είχατε ένα θέμα διαδικαστικό να θίξετε. Όχι. Ναι ή όχι. Όχι. Ωραία. Α, ναι. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να σας παρακαλέσω η 143 τροπολογία που αναφέρει κάποιες βραχυπρόθεσμες δυνατότητες ελέγχου μετά από συμφωνία δύο συγκεκριμένων κρατών, παραδείγματο χάρη για την αντιμετώπιση, αν θέλετε, ε, κάποιων ε, παράνομων δραστηριοτήτων, λαθρεμπόριων ναρκωτικών κτλ. Σε περιπτώσεις δύο κρατών που βρίσκονται σε συμφωνία, σε συνεργασία. Αυτό έχει προκύψει και με την Τσεχία. Για πολύ βραχυπρόθεσμες διάρκειες. Αφήστε με παρακαλώ πολύ να μιλήσω, συνάδελφοι. Ίσως μπορείτε να είστε ευγενεί, να με ακούσετε και μετά να αντιδράσετε. Αυτό που λέει η κυρία Χολμάιερ είναι ότι θα ήθελε να ψηφίσουμε ξεχωριστά. Αυτό λέει. Οκ, okay, όταν φτάσουμε εκεί, μπορείτε να το δεχτείτε. Απευθύνομαι στην εισηγήτρια. Η εισηγήτρια είναι εντάξει. Ναι, θα ψηφίσουμε λοιπόν ξεχωριστά για την τροπολογία αυτή. Όταν φτάσουμε στο σημείο αυτό. Is that okay, colleagues? Εντάξει, συνάδελφοι. Πάμε στην 25. Συμβαστική 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Okay, so the EPP have one... Έχουμε μία περισσότερη ψήφο από το ΕΛΚ. Πάλι αρχίσαμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. That is also carried. Εγκρίνεται. 143. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι ακριβώ πριν από την συμβαστική 24 στην σελίδα 4. 100 είναι η τροπολογία 143. Είναι αυτό που είχε ζητήσει προηγούμενα, ε, για ξεχωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν ξεχωριστά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 143 παρακαλώ. Ε, εξακολουθεί να είναι ανοιχτή η ψηφοφορία. Πέρα vote is closed. Απορρίπτεται. Συμβαστική 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Εγκρίνεται. Τροπολογία 146. Άρχεται η ψηφοφορία. 146. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τοπολογία 21 και 148. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 150 και 23 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 26 162 τροπολογίες, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 164 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 165 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21 Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Συμβαστική 20. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Μιλάμε για την συμβιβαστική τροπολογία 20. Ναι, 20. Α, είχα δίκιο. Ναι, είναι και τα γενέθλιά μου, γι' αυτό να είστε καλοί μαζί μου. Δεν ήθελα να με χειροκροτήσει, απλά είπα να με, να με φροντίζετε. Η συμβιβαστική 20, δεν έχουμε κλείσει ακόμα την ψηφοφορία, εγκρίνεται. Συμβαστική 21, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τι έγινε. Εγκρίθηκε η συμβαστική 21. Συμβιβαστική τρομολογία 22, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 185, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 23, ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 40 και 205 οι ταυτόσημες τροπολογίες, άρχεται η ψηφοφορία. 40 και 205. Αυτές εγκρίθηκαν ήδη, εντάξει, πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνονται. Τώρα έχουμε τις αιτιολογικές 43, άρχεται η ψηφοφορία. is Πέρας της ψηφοφορίας. Ε, απορρίπτεται. Ε, Τελογικές σκέψεις. Ε, συμβαστική 1. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Είμαστε στη συμβαστική 5, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τοπολογία 6, με συγχωρείτε. Ε, πρέπει να κάνουμε την τοπολογία 69, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 70 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 76 άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. εγκρίνεται 77 άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 78 άρχεται ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται και η τροπολογία 79 ξεκινάει η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 84 άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8 άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η ε, τροπολογία 91, άρχεται η ψηφοφορία. Με συγχωρείτε. Είναι η τροπολογία, δεν είναι συμβαστική, είναι τροπολογία 91. Έχω κουραστεί, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τι κάνουμε με την 95. Περνάμε στην συμβαστική 10. Ξεκινάμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έχουμε τροπολογία 103. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 115. Άρχεται η ψηφοφορία. Η τροπολογία 115. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα ε, ψηφίζουμε για το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί ε, διανομαστικής ψηφοφορίας. Άρχεται ψηφοφορία. Έχετε ψηφίσει όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 30, ε, έναντι 13. Ε, για την απόφαση να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Ναι. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 30, 24 κατά, χωρίς αποχές. Θα πάει στην Ολομέλεια αυτή έκθεση. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Έχουμε κλείσει την ψηφοφορία. Έχουμε μόνο ένα ακόμα θέμα στην μερισιά διάταξη. Thomas, non libe members will understand. Thank you, Thomas. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so um, colleagues, uh, we're going to move straight to. Συνάδελφοι, να περάσουμε αμέσω στο επόμενο σημείο. Είναι ο Ευρωπαϊκός Κωδικός για τις Θεωρήσεις. Να φύγουν, παρακαλώ, είναι να φύγουν για να ξεκινήσουμε εδώ τη συζήτηση με τους εισηγητές. Συνάδελφοι, εδώ έχουμε την παρουσίαση από τον εισηγητή, τον, Χουαν, τον, τον κ. Λόπεθ Αγγιλάρ, για τον κοινοτικό κώδικα θεωρήσεων που καθορίζει τους κανόνες, τους κανόνες για την έκδοση θεωρήσεων ε, μικρής διάρκειας ε, σε περίπτωση τράζιτ σε κάποιο αεροδρόμιο. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, στη συνέχεια στους κοινότητες εισηγητές και σε οποιοδήποτε άλλο μέλος θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά, συνάδελφοι, ε, που παραστήκατε στη συνεδρίαση τόσο αργά, μια Δευτέρα. Χωάν Φερνάντο, συγγνώμη και για το θόρυβο, σιγά σιγά θα ερεμήσουν τα πράγματα. Μπορείς να πάρεις το λόγο για να μας παρουσιάσεις το σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χρόνια πολλά, έστω και αργά απόψε, χρόνια πολλά. πολλά συγχαρητήρια. Κρατάω τα ακουστικά ακριβώς για να μην ακούω τον θόρυβο. Ε, θα είμαι σύντομος πάντως τους ή άλλως, μιας και είναι, παρότι, παρότι μάλλον είναι σημαντικό το ζήτημα, είναι καθήκον μου να παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης. Ε, δεν πρόκειται για κάποιο καινούριο θέμα κώδικα θεωρήσεων. Υπήρχε μια πρώτη πρωτοβουλία ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τη Δευτέρα το 2014 μάλλον είχε υποβάλει την πρώτη, είχε κάνει την πρώτη πρωτοβουλία, την απέσυρε τελικά και ήρθε με μια νέα πρωτοβουλία. Και αυτό είναι το σχέδιο έκθεση, τώρα το δικό μα. Το αποτέλεσμα ε, μια ε, σε βάθο προπαρασκευαστική δουλειά. Οι σκιώδεις συγητέ, τα άλλα μέλη συνεισέφεραν μετά από πρόταση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στις 20 Ιουνίου είχαμε και μια δημόσια ακρόαση ε, και για τις ανθρωπιστικές ε, θεωρήσεις και για τον κώδικα θεωρήσεων. Ε, τον Ιούλιο αυτή η ακρόαση συμμετείχαν πολύ ενδιαφερόμενοι, έγιναν πολλές συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς με την, και με τους και με μη οργανώσει, με προσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με άτομα, με πολίτε που εξέφρασαν ανησυχίε για το ζήτημα του υπάρχοντο κώδικα θεωρήσεων. Το σημείο αφιτηρία λοιπόν είναι ότι υπάρχει καλή θέληση για συμβιβασμό, να φτάσουμε δηλαδή σε μια συμβαστική λύση, υπάρχει ένα πνεύμα συμβιβασμού, να βρούμε μια κοινή θέση του Κοινοβουλίου ε, στη διαπραγματεύση με το Συμβούλιο. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο για να προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία. Νομίζω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει ε, να συνεργαστεί έτσι ώστε ε, έγκαιρα πριν από το τέλος δηλαδή αυτής της θητείας ε, να έχουμε ολοκληρώσει. Για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να εργαστούμε δυναμικά ε, όσο καλύτερα μπορεί ο καθένας. Θα έχουμε έναν πρώτο τρίλογο πριν από το Χριστούγεννα. Πριν δηλαδή το τέλος ε, της χρονιάς. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποια σχόλια για την πρόταση και για τις τροπολογίες ε, στο σχέδιο έκθεσης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου είναι τεχνικής φύσεως. Είναι εξαιρετικά τεχνικό. Ε, πρέπει να εξεταστούν αυτά τα τεχνικά ζητήματα λεπτομερώς τα κράτη-μέλη που είναι αρμόδια ε, για την εξέταση της, του αιτήματο, τα ταξιδιωτικά έγγραφα, τα υποστηρικτικά έγγραφα, για να μπορέσουμε να έχουμε υψηλά, ψηλές προδιαγραφές για να ε, ε, διασφαλίσουμε την δημόσια ασφάλεια και να, και να προστατευτούμε από την παραμετανάστευση, θα πρέπει να διευκολύνουμε το ταξίδι στους ταξιδιώτες ε, οι οποίοι είναι καλή την πίστη, bona fide. Θέλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε τα επίπεδα ασφάλειας, αλλά το νόμιμο, τους νόμιμους ταξιδιώτες, ε, τους νόμιμα ε, μετακινούμενους, να μπορούμε να στευκολύνουμε το έργο. Παίζει ένα κρίσιμο ρόλο αυτή η διαδικασία για τον κώδικα θεωρήσεων και σε οικονομικό επίπεδο. Γι' αυτό είχαμε και επισκέψεις οικονομικών παραγόντων. Ο τουρισμός, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ σημαντικός για κάποιες περιοχές, όπως η δική μου. Και η δυνατότητα λοιπόν του να μπορεί κάποιος ηλεκτρονικά να συμπληρώνει τις αιτήσει. Ε, υπάρχουν λοιπόν κάποια τεχνικά στοιχεία στο κείμενο. Η διευκόλυνση πάντως είναι στην καρδιά αυτής της πρωτοβουλίας. Η απλοποίηση. Η παρούσα πρόσθεση τη Κομισιόν συνδέει την πολιτική θεωρήσεων με την εξασφάλιση μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των ζητημάτων μετανάστευση και των ζητημάτων ασφάλεια. Τα οικονομικά ζητήματα, γενικότερα τι εξωτερικέ σχέσει, μπαίνουν και πολιτικά ζητήματα. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ τη μετανάστευση και ασφάλεια αφενό και τη διευκόλυνση τη χορήγηση θεωρήσεων από την άλλη. Να μην δηλαδή μα πνίξουν τα ζητήματα ασφαλεία, Αυτό είναι που με ανησυχεί εμένα. Επίση, δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως άλλωστε είπε και η, αρχή, η Εποπτική Αρχή προστασία Δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Αρχή, επανειλημμένα αναφέρεται στη μετανάστευση για ζητήματα ασφάλειας, καταπολέμησης τρομοκρατίας, ε, ε, ότι δεν πρέπει όμω αυτό ε, να, το, να το ταυτίζουμε. Δεν πρέπει δηλαδή ε, να είναι συγκεκριμένε οι γραμμέ μεταξύ των απλών ταξιδιωτών και την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Θα πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό. Σε αυτό το σημείο ισορροπία μεταξύ ασφάλεια και ελευθερία και τη χρήση τη πολιτική θεώρηση για να πετύχουμε κάποιου πολιτικού στόχου, ε, υπάρχουν και τα οικονομικά ζητήματα, τα εξωτερικά ζητήματα, τα οποία όμω λείπουν στην πρόταση εάν το συγκρίνουμε δηλαδή με την πτυχή που φορά την ασφάλεια και που είναι πολύ πιο έντονη, θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε τόσο στο σημείο ισορροπία. Οι οικονομικέ πτυχέ που έχουν να κάνουν με του καλόπιστου ε, ε ταξιδιώτε και τα ζητήματα ασφάλεια. Επανειλημμένα, μελέτη δικτύπου τη Κομισιόν αναφέρεται στην αυξανόμενη μετανάστευση, του κινδύνου για την ασφάλεια. Ταυτόχρονα, ε, βεβαίω, ε, ε, παραδέχεται το, η μεγάλη πλειοψηφία των ετούντων θεώρησης δεν δημιουργούν κανένα ζήτημα ασφάλειας. Δεν θέλουν να μεταναστεύσουν. Θέλουν να μπουν στο έδαφος της Ένωσης για έναν καλό σκοπό. Η πρόταση αυτή λοιπόν δεν είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη, είναι απαραίτητο στις διαπραγματεύσει και με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο να βρεθεί το σωστό σημείο ισορροπία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και την άποψή μα. Θα θυμάστε ότι υπήρχε πρόθεση να συνδέσουμε το κώδικα θεωρήσεων με το να ανοίξουμε ένα νόμιμο, μια νόμιμη οδό, ανθρωπιστικές θεωρήσεις, ε, ε θεωρήσεις ε, για ευάλωτες ομάδες. Τελικά δεν μπόρεσε να προχωρήσει αυτό. Έφυγαν, έφυγε οποιαδήποτε αναφορά στα ζητήματα αυτά. Ε, ευτυχώς ε, η πλειοψηφία της Επιτροπής Λίμπε τα είχε εγκρίνει αυτά και ελπίζω η Ολομέλεια αυτό ε, να το επιβεβαιώσει τον Νοέμβριο και να στείλουμε ένα μήνυμα για να δημιουργηθεί πρόοδος γρήγορη, ε, επικεντρωνόμενη στο περιεχόμενο της παρούσας πρότασης ε, ξεχωριστά, μόνο δηλαδή τον κώδικα θεωρήσεων. Το πιο λεπτό ζήτημα για μένα είναι ο νέος ρόλος για την πολιτική θεωρήσεων ως μοχλός για την πολιτική επανεισδοχής συμφωνίες επανεισδοχή. ε, αναφέρεται αυτό σε πολλά έγγραφα, ότι πρέπει να έχουμε κατά νου και τα ζητήματα επανεισδοχή. Όμω είναι η πρώτη φορά που ενσωματώνεται κάτι τέτοιο σε ένα νομοθετικό κείμενο. Συνδέουμε την χορήγηση θεώρηση με τι συμφωνίες επανεισδοχή με τρίτε χώρε ό,τι αφορά του παράτυπου μετανάστε. Ε, η Κομισιόν βεβαίω παραδέχεται ότι αρχικά ο κώδικα θεωρήσεων δεν είχε αυτό το σκοπό να είναι δηλαδή ένα ε, μοχλο πίεση για τι τρίτε χώρε για να δεχθούν συμφωνίε πανεσδοχής. Θέλαμε απλώ να ευθυγραμμίσουμε τις διαδικασίες χορήγησης θεώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά όμω, ε, με αυτό το νέο πολιτικό πλαίσιο όπου υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία για τα ζητήματα ασφάλεια, αλλάξαν τα πράγματα. Επίση, αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι σαφέ ότι καλύτερη συνεργασία για ζητήματα πανεσδοχή με τρίτε χώρε οι οποίε διστάζουν δεν πρέπει να επιτευχθεί μόνο μέσω της πολιτικής θεωρήσεων. Ε, θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα πολιτικό μείγμα με θετικά κίνητρα, αντικίνητρα ε, στον τομέα της ανάπτυξης, ε, της συνεργασίας, της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, της οικονομικής συνδρομής. Ε, αυτή, αυτό το πολιτικό μείγμα όμως δεν είναι και τόσο εμφανές αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει επίση μια έλλειψη δεδομένων, στοιχείων. Στην ε, αξιολόγηση αντικτύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ρητά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το πώς μπορεί αυτή η πίεση σε ζητήματα θεώρησης θα βοηθήσει ε, στη συμφωνία επανεισδοχής με τρίτες χώρες. Ε, με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Θα πρέπει πραγματικά να πούμε ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα την, την μελέτη αντικτύπου της Κομισιόν. Αυτό το θέμα δηλαδή της αύξησης της, ε, των μοχλών πίεσης ε, δεν αναλύεται συγκεκριμένα. Χρειάζονται δηλαδή πολύ πιο συγκεκριμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν το σχετισμό. Τέλος, υπάρχει εδώ κάτι το παράδοξο. Και το Συμβούλιο και η Κομισιόν ε, λένε ότι δεν πρέπει εδώ στα ζητήματα ε, ε, θεώρησης, κώδικα θεωρήσεων να μιλήσουμε για ανθρωπιστικέ θεωρήσεις, δεν έχει θέση εδώ αυτό, αλλά θέλει να το χρησιμοποιήσει όμω ε, τι θεωρήσει για τις εμφανίσεις πανεσδοχής. Ε, λοιπόν, πρέπει να βρεθεί ένα σημείο ισορροπία με σχέση με την πρόταση τη Κομισιόν για να την βελτιώσουμε. Το δεύτερο είναι η ε, ιατρική ασφάλιση. Δεν πρέπει να ζητείτε από τους ταξιδιώτες να προσκομίζουν έγγραφα περίπλοκα ε, ιατρική ασφάλιση όταν ζητούν μια θεώρηση μια σύντομη, ε, για μια σύντομη διαμονή. Ε, είναι ένα δυσανάλογο βάρο αυτό για τους ετούντες θεώρηση. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία, κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι οι κάτοχοι θεώρηση μικρή διάρκεια αποτελούν κίνδυνο για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν εδώ μια τροπολογία για να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Τώρα, το τρίτο σημείο, η γενικότερα διαδικασία χορήγηση θεώρηση. Ε, πρέπει να ενισχυθεί η πρόταση. Θα πρέπει να μπορεί κάποιο να υποβάλει την αίτηση όχι μόνο έξι μήνε πριν ε, το ταξίδι, αλλά και εννέα μήνε Για να μπορεί ε, να ταιριάζει και με ε, τον, χρόνο των πιο φτηνών εισιτήριων. Ε, όσο πιο νωρίς αγορές τόσο το καλύτερο. Υπάρχει το, το θέμα των πολλαπλών ε, θεωρήσεων, ε, χωρίς θεωρήσεις πολλαπλών, πολλαπλών εισόδων. Είναι ένα πλεονέκτημα αυτό, όχι μόνο για τους καλόπιστους, τους bona fide ε, ταξιδιώτες, αλλά και για τα προξενία. θα υποβάλουμε λοιπόν τροπολογίες για να βελτιωθεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Συνεχίζει όμως ο κ. Λόπε Αγγιλάρ, ε, τα περισσότερα προξενία ήδη έχουν κάποιε βέλτιστε πρακτικέ ε, και επίση βεβαίω όταν υπάρχει άρνηση χορήγηση θεώρηση πρέπει να υπάρχει κάποια δυνατότητα προσφυγή ε, για, τον, του ενδιαφερόμενου. Στα προξενία και κλείνω λέγοντα ότι είμαστε στην αρχή τη διαπραγμάτευση και με μονησία την συνεργασία σε ένα επικοδομητικό πνεύμα. Ναι, αφήστε τα καλύτερα για αργότερα. Ε, δεν ξέρω αν θέλω να πω κάτι σκιώδεις εισηγητές, σύντομα όμως. Εντάξει, ο Χάιντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτή την πρώτη παρουσίαση που μας κάνει. Διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για απλούστευση της διαδικασίας, δίνονται θεωρήσεις σε άτομα από τρίτες χώρες με σκοπό να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας για καλλιτέχνες, για αθλητές, για τουρίστες, για επιχειρηματίες. Αυτός είναι ο σκοπός. Και βεβαίως το θέμα της ανθρωπιστικής βίζας. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεχωριστό πακέτο, ξεχωριστός φάκελος. Και εδώ βρήκαμε βέβαια μια συμβαστική λύση με τον εισηγητή και το ολο, ολοκληρώσαμε. Αλλά εδώ σε αυτή την έκθεση βλέπω προσπάθειες να ενσωματωθεί κάπως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό το θέμα των ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Θα ζητήσουμε μέσω τροπολογιών ξεχωριστή ψηφοφορία. Το θέμα της επανεισδοχής και των επιστροφών. Ναι, βεβαίως αυτό εδώ πρέπει να ενσωματωθεί. Γιατί, γιατί αφού την ε, διεκπαιρέωση των θεωρήσεων για τις τρίτες χώρες αυτές θα πρέπει και δείχνουμε καλή πίστη και καλή θέληση, θα πρέπει και οι τρίτες χώρες αυτές σε περιπτώσεις προβλημάτων να μπορούν να δεχτούν τους υπηκόους τους με έναν απλό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, το θέμα των ασθενών οι οποίοι αν θέλετε επισκέπτονται τη μία ή την άλλη χώρα και οι οποίες κάποιες φορές πρέπει να δοθούν θεωρήσεις. Πιστεύω ότι θα ασχοληθούμε με πολλές τροπολογίες. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες επιπλέον και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην δίνουμε φανταστικές ελπίδες και προσδοκίες, αλλά να είμαστε ρεαλιστές, να το προσπαθήσουμε τουλάχιστον και αυτό να ενσωματωθεί στις τροπολογίες μας, αλλιώς θα αποφασίσει η ψηφοφορία. Πρόεδρος, να είσαστε σκιώδης για την ICR. έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ προσεκτικά διάβασα την έκθεση και ήδη είπα και επαναλαμβάνω ότι άλλο είναι οι θεωρήσεις και άλλο οι επιστροφές, αλλά υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των δύο. Αν μια χώρα δεν δέχεται να επιστρέψει και να δεχθεί έναν ε, υπήκο της χώρας αυτής, ο οποίος έχει εγκατασταθεί παράνομα στη χώρα μας, γιατί να προσφέρουμε εμείς ελαφρύνσεις όσον αφορά τη διαδικασία των θεωρήσεων. Πραγματικά εκπλήσωμα γιατί εδώ ο εισηγητής θέλει να παραλείψει τις προτάσεις αυτές και τα άρθρα αυτά που ξέρουμε ότι είναι απαραίτητα για να υπάρξει συμφωνία του Συμβουλίου. Δεν θέλουμε να ενσωματωθούν, παραδείγματος χάρη, πολιτικά θέματα στον ε, κώδικα για τις θεωρήσεις. Ναι, βεβαίως. Για θέματα επενδύσεων, για θέματα κοινωνικά, για θέματα εκπαιδευτικά. Εδώ μιλάμε για ελάφρυνση των θεωρήσεων. Το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Και πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, να υιοθετηθεί το θέμα αυτό πριν τις επόμενες ε, εκλογές. Και είναι πολύ κρίμα, πραγματικά απαράδεκτο, γιατί σκοπός μας είναι να διευκολύνουμε τις μετακινήσεις και τον τουρισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Αυτός ο, ο κώδικας ήταν το πρώτο θέμα που έφτασε στο γραφείο μου όταν ήρθα το 2014 στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχαμε μια πρόταση από την Κομισιόν τότε που χρησιμοποιούσαμε για να βασίσουμε τη δουλειά μας, όπως γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχουν πάντα προβλήματα που προκύπτουν, για παράδειγμα όταν δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για την ανθρωπιστική θεώρηση. Ακόμη και αν στο παρελθόν πολλές φορές είχαμε συμφωνήσει ότι οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε. Είναι κρίμα που ακούμε ότι αυτή η συνοχή που είχαμε κάποτε, μια φορά και έναν καιρό, στα θέματα ανθρωπιστικών θεωρήσεων, έχει τώρα ε, μειωθεί και ε, ο κωδικός που συζητούσαμε τότε ε, ως μέσο διευκόλυνσης των ατόμων που μας επισκέπτονται για διάφορους λόγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν ένα θέμα διευκόλυνσης, όχι, ε, δεν, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πιο δύσκολη τη ζωή των ανθρώπων. Τώρα έχουμε ένα νέο κώδικα που αντί να διευκολύνει ε, βάζει εμπόδια ε, στο δρόμο των ανθρώπων. Αν και υπάρχουν πλέον εκτήματα, υπάρχουν όμως περισσότερα μείον εκτήματα. Για παράδειγμα, κάτι που ήδη αναφέρθηκε σχετικά με τις συμφωνίες επανεισδοχής. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη, αυτό το συγκεκριμένο κώδικα ε, υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτό. Υπάρχουν άλλοι τομείς που το εξετάζουμε και ε, πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να το αφήσουμε έξω από τον κώδικα θεωρήσεων, όπως και αυτό που είπαμε, για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις, ότι δεν πρέπει να περιληφθούν. Γιατί πρέπει να περιληφθεί αυτό το θέμα της επανεισδοχής. Τα περισσότερα πράγματα τα έχουν αναφέρει οι προηγούμενοι. Ωστόσο θέλω να κάνω ένα σχόλιο και να επανέλθω στην ανθρωπιστική ε, θεώρηση. Έχουμε ψηφίσει ε, μια πρόταση για ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Άρα έχουμε διανύσει ένα μέρος του δρόμου, όμως έχουμε ακόμη μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Εάν είναι εθελούσια ε, εφαρμογή για τη χρήση της ανθρωπιστικής θεωρήσης, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Και έχουμε και πολύ, ε, πολύ απόσταση μεταξύ μας εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Στα περισσότερα σημεία συμφωνώ ε, για τον κώδικα των θεωρήσεων. Ευχαριστώ, Μαρή Κριστίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καμιά φορά να ρωτιέμαι πραγματικά ποιο είναι το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε εδώ. Νομίζω ότι έχω, παρατηρεί, έχω παρακολουθήσει το θέμα από την αρχή. Ο κώδικας θεωρήσεων και η μεταρρύθμιση του, η ανθεώρησή του, είχε σαν σκοπό τη διευκόλυνση των τουριστών. Εδώ ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι έχει μετατραπεί σε ένα εργαλείο για την καταπολέμηση της παράνομης ή λεγόμενης παράτυπης μετανάστευσης. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που κάθε χρόνο εκδίδει περίπου το 1 τέταρτο των θεωρήσεων. Ε, θα πρέπει λοιπόν λίγο να ξανασκεφτούμε αυτό το θέμα, διότι εδώ μπαίνουν εμπόδια και περιορισμοί που δεν έχουν καμιά σχέση με τις ε, θεωρήσεις ε, μικρής διάρκειας. Δεν έχει καμία σχέση το θέμα αυτό. Ουσιαστικά ο Ευρωπαίος πολίτης δεν έχει καμία, αν θέλετε, τέτοιου είδους ανησυχία. Θέλει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα, να μπορεί να υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία και διαπιστώνω ότι αυτός ο κώδικας θεωρήσεων ουσιαστικά εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταγμά. Δηλαδή εμείς που έχουμε τη δυνατότητα και την τύχη να ζούμε και να έχουμε γεννηθεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα, έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες και ελευθερία να κινηθούμε στον κόσμο σε σχέση με τους υπηκόους τρίτων χωρών. Δεν καταλαβαίνω γιατί ουσιαστικά εξαρτάται η δική μας στάση και το αν ναι ή όχι θα δοθεί βίζα σε κάποιον από τη στάση της κυβέρνησης της εν λόγω χώρας. Όσον αφορά τα Εμμυράτα, παραδείγματο χάρη, έχουμε απελευθερώσει τις θεωρήσεις ε, για τις χώρες αυτές. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο για την επικαιρότητα, αλλά πραγματικά πως πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Εγώ διαφωνώ όσον αφορά το θέμα της σύνδεσης του θέματος αυτού με το θέμα της επανεισδοχής και της επιστροφής. Μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό, για το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία για τους υπηκόους αυτών των χωρών. Και δεν πρέπει να το συνδέσουμε αυτό με τίποτα άλλο. Δεν πρέπει να βάλουμε όρους και προϋποθέσεις. Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή όσον αφορά την ανθρωπιστική θεώρηση. Δεν έχει καμία σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αναφερόμαστε στο δικαίωμα κάποιων ανθρώπων των οποίων απειλείται η ζωή να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Σιγητά, σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με τις περισσότερες προτάσεις σας θα επιμείνω σε αυτά με τα οποία έχω δυσκολία. Είμαι κατά της αύξησης της τιμής των θεωρήσεων. Γιατί, γιατί σιγά σιγά θα γίνει εργαλείο για τους πιο πλούσιους και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν τα προξενία να ζητήσουν να πληρωθεί, αν θέλετε, αυτή η πολιτική ανάθεση σε εξωτερικούς φορείς, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Και αυτό που συμβαίνει είναι σε πολύ φτωχές χώρες όπως την Ιπποσαχαρία Αφρική οι βίζες να στοιχίζουν εξαιρετικά ακριβά. Επίσης, το θέμα της υγείας. Και εκεί δεν συμφωνώ με τον εισηγητή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο τολμηροί όσον αφορά παραδείγματο χάρη τις οικογενειακές σχέσεις και αυτόν παραδείγματο χάρη που θα υποδεχθεί κάποιον που φτάνει σαν τουρίστας στην Ευρώπη. Και εδώ είμαστε λίγο υπερβολικοί και είναι παράλογες οι προτάσεις αυτές που κάνουμε. Επιθυμώ, αν και ξέρω ότι έχουν γίνει προτάσεις και από τον εισηγητή και από την Επιτροπή, δεν καταλαβαίνω γιατί περιορίζουμε τους εκπροσώπους οργανώσεων, συλλόγων που επισκέπτονται τη χώρα για λόγους συμμετοχή σε κάποια σεμινάρια. Γιατί βάζουμε όριο ηλικία. Πολλέ φορές οι χώρε αυτέ εκπροσωπούνται από πιο ηλικιωμένα άτομα. Δεν είναι μόνο για τους νέου αυτά τα ταξίδια. Κύριε Σιγητά, θα υποβάλω κάποιε τροπολογίες βάσει αυτών που σας παρουσίασα και ελπίζω να έχουμε καλή συνεργασία μεταξύ μας γιατί σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με το πνεύμα των ε, προτάσεών σας. Um, Ευχαριστώ Μαρή Κριστίν. Ε, ουσιαστικές οι συνεισφορές των σχεδόν εισηγητών ε, αλλά και από τον εισηγητή. Λοιπόν, θα σταματήσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Ε, 5 Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Σα ευχαριστώ συνάδελφοι και για την υπομονή σα. Ξέρω ότι είναι πολύ αργά. Βλέπω ότι είναι εδώ και ο Τέρι Κάβερ. Να πάμε στο επόμενο σημείο κατευθείαν. Είναι και σκιώδεις ηγητέ εδώ. Σας, θέλω να σα ευχαριστήσω όλου ε, για την υπομονή σα και για την αντοχή σα. Πάμε απευθεία λοιπόν στο ζήτημα τη κατάσταση των θεμελιών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2017, σχετική έκθεση. 6 Σεπτεμβρίου ο κ. Τέρι Κάμπρα, ε, ο εισηγητή για αυτή την έκθεση, υπέβαλε το σχέδιο έκθεση με πάνω από 400 τροπολογίε. Ε, θα μας ε, παρουσιάσει τώρα αυτές τις τροπολογίες περιμένει με μεγάλη υπομονή ο κ. Κάμπρας εδώ και πολλή ώρα. Ε, είναι και δύο σκέδες συγκίτες εδώ. Έχετε το λόγο να, να συγχαρώ πραγματικά και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έκατσαν μέχρι τόσο αργά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος, διότι είναι αργά και είμαστε κουρασμένοι. Και πρέπει και εσείς κάπου να γιορτάσετε τα γενέθλιά σας. Ε, ιδιωτικά, φαντάζομαι. Ναι, απλώ να ξαναπούμε ότι είναι τα γενέθλιά μου, έτσι, διότι κάποιοι ενταχώ να μην το ξέρουν και κοιτάζουν, με κοιτάζουν απορριμμένοι. Ε, θα ήθελα λοιπόν πρώτα να ευχαριστήσω του σκιώδει συγγενεί για το έργο του ε, στην έκθεση αυτή για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όπω είπατε, είχαμε 460 τροπολογίες ε, που θα εμπλουτίσουν το τελικό κείμενο. Θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι έχουμε λιγότερες τροπολογίες από ότι τα προηγούμενα έτη. Αυτό βεβαίω μπορεί να ερμηνεύσει κανεί με διάφορου τρόπου. Ε, είναι καλό σημάδι, θα έλεγα πάντω. Οι σκιώδει ηγητέ ε, δηλαδή συμφώνησαν με την ιδέα ότι πρέπει να είμαστε ε, συνεκτικοί. Εξετάζοντα τι τροπολογίε, ε, διαπίστωσα ότι έχουμε μια κοινή προσέγγιση για το γενικότερο περιεχόμενο ε, σε ό,τι αφορά τη θεμελιώδη δικαιώματα πέρυσι. Ε, η ελευθερία του τύπου, ε, LGBTI, προστασία των whistleblowers, ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία των μειονοτήτων και βεβαίως η αύξηση των ακροδεξιών κινημάτων. Ένα από, ένας από τους βασικούς στόχους μου σε αυτή την έκθεση είναι να εντοπίσουμε ποια είναι τα, τα ζητήματα εκείνα που, είναι στο που ήταν στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ζωής το 2017, χωρίς καμία πρόθεση βεβαίως να ε, παραμελήσουμε το οτιδήποτε. Επελέγησαν αυτές, ε, αυτά τα ζητήματα λόγω του πολιτικού κοινωνικού αντικτύπου και λόγω του επίγοντος ε, των ζητημάτων αυτών. Όπως είπε, είπαμε και με mail στην γραμματεία της ΛΥΜΠΕ, 19 Οκτωβρίου θα έχετε το κείμενο σε όλες τις γλώσσες. Η πρώτη συνάντηση των σχεδόν εισαγητών θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου 10 με 11 και μισή. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλους τους σκιώδες εισηγητές για, αυτό για αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τερικάμπρας. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική η έκθεση για δικαιώματα. Πάντα υπάρχουν πάρα πολλέ τροπολογίε. Ε, αυτό σημαίνει πολλή δουλειά. Η Σιλβή έχει το λόγο και η συγκεντρία για του Σοσιαλιστικού Δημοκράτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω τον Τέρι που ανέφερε όλα αυτά που ανέφερε. Τηλεγραφικά όλα θα πάνε πολύ καλά εάν ε, ξισορροπήσουμε ε, τα διάφορα ζητήματα. Το έχουμε ξαναπεί ότι τα ζητήματα κράτους δικαίου είναι πολύ σημαντικά, είναι στην πρώτη θέση, νομίζω εκεί δεν θα υπάρξει θέμα και όλα θα πάνε καλά επίσης εάν ε, συμφωνήσουμε για το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών. Ε, το λέω έτσι αυτό, ε, το αναφέρω, μην το ξεχνάμε, δίνοντας έμφαση στο θέμα ε, της ε, παρενόχλησης, των εγκλημάτων μίσους επίσης, υπάρχουν πολλά θέματα εδώ για τα ε, δικαιώματα της, των μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, ε, των Ρωμά, ε, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα μετάσταση και ασύλου, επίσης σημασία της προστασίας των μελών δικαιωμάτων, διότι υπάρχουν παράνομες πρακτικές σε πολλά κρατημέλη και τέλος έχουμε και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων, των fake news. ελπίζω λοιπόν να τα βρούμε ε, και ελπίζω να καταφέρεις τέρι να ε, καταργήσεις ε, ε, μια σειρά από τροπολογίες εξαιρετικά δύσοσμες, ιδιαίτερα για τα δικαιώματα των γυναικών και την βία, πραγματικά ξεπερνούν και το παράλογο αυτές τις τροπολογίες. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο τέτοια ώρα κιόλα. Είναι η στιγμή όμως που, τη ημέρα, έτσι αργά το βράδυ, που είμαστε και πιο ειλικρινεί. Πάντω δεν θέλω να έχουμε άλλε τέτοιε συναντήσει τέτοια ώρα. Ε, Μαρή Κριστίν, ε, υπάρχει κάποιο θέμα που να μην είσαι και όχι γητριά. Νομίζω πω θα έπρεπε ε, να είσαι στην πρώτη, στην πρώτη θέση βαθμολογία για του πιο σκληρά εργαζόμενου ε, ευρωβουλευτέ. Σε χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Πρόεδρε, θέλω να σα πω. Ναι, πολύ σύντομα, διότι δεν έχω καμιά διαφωνία ούτε με τον ε, εισηγητή, ούτε με αυτά που είπε Έχουμε τις ίδιες ανησυχίες ε, σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Νομίζω όμως ότι μας ακούσατε από αυτού και ότι όντως ε, πρέπει να αρχίσουμε από αυτό. Μεταξύ των ανησυχιών των πιο προσωπικών ή της ομάδας μου, όπως περιπτώσει, ε, έχουμε το θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ε, της, του σεβασμού των θεμελιών δικαιωμάτων, το δικαίωμα ασφάλειας των πολιτών βεβαίως δεν πρέπει ε, να πλήττει τα θεμελιώδη δικαιώματα, να αποφύγουμε επίσης το να τσουβαλιάζουμε τη μετανάστευση, την τρομοκρατία και την εγκληματικότητα. Δεν θέλω και εδώ τώρα να πω τι λένε άλλοι για αυτά έχω και μια ανησυχία για το θέμα της αστυνομικής βίας. Καλό θα ήταν και αυτό το ζήτημα να ενσωματωθεί. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό αυτά που είπε η Σιλβή για το θέμα της καταπολέμησης των διακρίσεων. Επειδή είναι αργά, δεν θα πω κάτι περισσότερο από αυτού. Επίσης, υποστηρίζω τον εισηγητή στο αίτημά του, στην βούλησή του, να πάει λίγο παραπέρα στην ανάγκη υποστήριξης της υπηρεσίας των δικαιωμάτων. Για άλλη μια φορά, χρόνια πολλά, Πρόεδρε. Ε, προηγουμένως ενδεχομένως να μακρηγόρησα, τώρα όμως ε, σας τα δώσα πίσω. Ευχαριστώ. Και Γιούρεκ, ε, με συγχωρείτε, δεν είχα προσέξει ότι ήσασταν εκεί. Δεν ξέρω γιατί κάθεστε τόσο μακριά. Είστε ο Σκιώδης ε, από πλευρά CCR για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ και ε, να τα εκατοστήσεις που λέμε στα γενέθλιά σου. Αυτό για να ξεκινήσω. Θα ήθελα λοιπόν να σου ευχηθώ να τα εκατοστήσεις. Τώρα, σχετικά με την έκθεση, εμείς βλέπουμε ότι είναι κάπως μονόπλευρο το κείμενο. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ισορροπία του με τις τροπολογίες μας, ιδιαίτερα στο θέμα της ελευθερίας ε, της ανεξιθρησκείας μάλλον. Και αυτό δεν υπάρχει στο κείμενο, δεν αναφέρεται το κείμενο σε θέματα ε, επιθέσεων κατά ε, θρησκευτικού δόγματος. Ε, αυτές οι τροπολογίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα είναι μια πράξη καλής πίστης και θα οδηγήσει και σε μια πιο περιεκτική έκθεση σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα ήθελα επίση να φυστήσω την προσοχή σας στο γεγονό ότι δεν μιλάμε και για τα δικαιώματα των της οικογένειας. Για παράδειγμα, το δικαίωμα των γονιών να μορφώσουν, να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους. Αυτό αναφέρεται ρητά στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν αναφέρεται η χειραφέτηση ε, ε, ομάδων που, έχουν, ε, που τυχάνουν διακρίσεων, που έχουν ε, περάσει από ολοκληρωτικά καθεστώτα θα πρέπει να φαίνεται η πραγματική ε, κοινωνική ισότητα και αυτό δεν αναφέρεται στο κείμενο. Το κείμενο περιέχει κάποιες, ε, κάποια κενά. Βλέπουμε το άρθρο 7 και αναφερόμαστε σε αυτό που είναι σαφέστατο και είναι σαφές γιατί στήριζεται σε κάποια ξεκαθαρή φιλοσοφία. Ή ε, λέμε ότι το άρθρο 7 α, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ε, έναν μηχανισμό που δεν στηρίζεται στις συνθήκες και εδώ νομίζω ε, ξεφεύγουμε από τις συνθήκες με αυτή την ε, κίνηση. Πάνω από όλα λοιπόν θα θέλαμε να εισηγηθούμε ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και επίσης μαζί με όλους θα αναφέρω και εγώ την ανάγκη να λάβουμε υπόψη το θέμα της διαφθοράς. Η διαφθορά είναι μία πράξη ε, αδικίας, μη δικαιοσύνης ε, σε ό,τι αφορά ε, άτομα που δεν μπορούν να έχουν ίσες αποφάσεις. Αλλά υπάρχουν χώρες όπου ακόμη και υψηλόβαθμοι οι αξιωματούχοι στη χώρα, στις αρχές της χώρας, επιδίδονται σε παράνομες ενέργειες. Ε, θα πρέπει να υποβάλουμε λοιπόν τις τροπολογίες μας και θα ήθελα να τις λάβετε υπόψη. Ευχαριστώ κύριε Γιούρεκ. Κύριε Τερικάπρας. Συμφωνείτε. Δεν σας βλέπω, αλλά θέλετε να πείτε κάποια καταληκτικά λόγια. Ναι. Να πω ότι ε, ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Ελπίζω να δουλέψουμε σε ένα επικοδομητικό πνεύμα και να πετύχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι. Το ελπίζω. Ευχαριστώ κύριε Τερικάπρας. Ε, νομίζω δεν θα μου το συγχωρέσετε ποτέ ότι έχουμε μια συνάντηση τώρα ε, τέτοια ώρα, 9 και 20. Έχουμε άλλο ένα θέμα όμως στην ημερησία διάταξη. Το 7. Εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης σχετικά με την ηθαγένεια. Δεν βλέπω όμως την εισηγήτρια στην αίθουσα ή μήπως υπάρχει αντικαταστάτη της. Δεν είναι εδώ ότι είναι αντικαταστάτρια. Ο κ. Σόκο, Σκιώδης είναι. Ήρθατε εδώ για αυτό το θέμα. Εκ μέρους ε, της, της συντάκτριας και της αντικαταστάτριας ε, που δεν βρίσκονται εδώ, δεν είναι και πολύ καλό γιατί οι σκιώδεις αφιέρωσαν τον χρόνο τους. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους τους, διότι είναι πάρα πολύ αργά και λυπάμαι πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Θα πρέπει να αναβάλουμε τη συζήτηση του θέματος Συγγνώμη λοιπόν προς τους δύο σκιώδεις που βρίσκονται εδώ. Um, I don't think that's conventional. Uh, Sylvie, just before you go, would you... πρωτού φύγεις, ε, απευθύνομαι στους σκιώδες. Θα θέλατε να μιλήσετε και να μιλήσουμε στη συνέχεια για τις προθεσμίες. an option if you want. Εάν θέλετε να έχετε το λόγο, είναι μια επιλογή που σας δίνουμε. Θέλετε να απευθύνετε το λόγο εδώ. Ό,τι θέλετε θα κάνω, αλλά βεβαίως εγώ μπορώ να αντικαταστήσω την κυρία Κέγκε, έχω ένα κείμενο, μπορώ να το διαβάσω, μπορώ να μην το διαβάσω, ό,τι θέλετε. Εγώ προτιμώ να το αναβάλουμε το σημείο αυτό. Ζητώ συγγνώμη στους δύο σκιώδεις που είναι παρόντες και ήρθαν για το σημείο αυτό, για τα μέλη, επίσης ζητώ συγγνώμη σε όλους το προσωπικό. Σας ευχαριστώ που με μεγάλη υπομονή ήσασταν παρόντες και περιμένατε. Τέλος της συνεδρίας.